με πολύτιμες ζωέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κλείνουμε τη συζήτηση αυτή και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12.30. Ε, Προχωρούμε τώρα σε ένα άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη ε, την έκθεση της κυρίας Ρόδης Κράτσα Τσαγκαροπούλου «Ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων στην Ευρώπη». Και καταρχήν θα δώσω το λόγο στην κυρία η συγγήτρια για τέσσερα λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, οι αποφάσεις των τελευταίων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη για την έξοδο από την δημοσιονομική και την οικονομική κρίση. Η ανάπτυξη αποτελεί το βασικό φάρμακο. Θα δημιουργήσει πλούτο, θέσεις εργασίας, θα συμβάλλει στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και θα ενισχύσει την οικονομική και την περιφερειακή σύγκληση. η ανάπτυξη θα προέλθει ε, κατεξοχήν από επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις. αυτό είναι το θέμα της έκθεσης που ε, συζητούμε απόψε πώς η ευρωπαϊκή ένωση θα έλξει ξένες επενδύσεις πώς θα ε, ενισχύσει το επιχειρηματικό πνεύμα των ίδιων των ευρωπαίων και θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να επενδύσουν οι ευρωπαίοι ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μέλη της επιτροπής οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων για τις πολύτιμες ιδέες τους που εμπλουτίζουν την έκθεσή μου και επίσης και τους συναδέλφους από τις άλλες επιτροπές που γνωμοδότησαν με πολύ στοχευμένες παρατηρήσεις. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλη τη σχετική κάμψη, παραμένει ο πρώτος επενδυτικός προορισμός στον κόσμο αλλά με δεδομένους τους κινδύνους που εγκυμονούν αφενός η δημοσιονομική κρίση που μας στερεί πόρους για επενδύσεις και αφετέρου η ανάδυση νέων ανταγωνιστικών επενδυτικών προορισμών πρέπει να μας κινητοποιήσουν για να προστατεύσουμε τη θέση της ένωσης. πρέπει να δράσουμε παράλληλα σε ευρωπαϊκό και σε τοπικό εθνικό επίπεδο. καταρχάς για την σταθερότητα τη δημοσιονομική ε, και την νομισματική, την ε, εμπιστοσύνη στις διεθνείς αγορές, αλλά και στους ίδιους τους Ευρωπαίους, τους επενδυτές και τους καταναλωτές. Πρέπει να θωρακίσουμε το τραπεζικό μας σύστημα για να μπορέσουμε να έχουμε ρευστότητα στην αγορά, αποτελεί το βασικό μοχλό για τις επενδύσεις η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να επενδύσει στα πλεονεκτήματά της. χρειαζόμαστε δημόσιες και ιδιωτικέ επενδύσεις και στοχευμένες κοινωνικέ επενδύσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου που αποτελεί από τα βασικά πλεονεκτήματα της ένωσης. να ενισχύσουμε την ενιαία αγορά τι διασυνοριακέ ε, συνεργασίε ε, και τον εξυγχρονισμό της ε, αγορά δημοσίων συμβάσεων να αναπτύξουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα να αξιοποιήσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία για να δώσουμε τη δυνατότητα επενδυτικής ελκυστικότητας σε όλες τις περιοχές ανάλογα με τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. σε διεθνές επίπεδο η ένωση πρέπει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για πολυμερείς ε, ή διμερείς συμφωνίες ε, που θα δώσει ωφέλη στο εμπόριο και στις επενδύσεις για την ίδια την ένωση και επίσης σε διεθνές επίπεδο πρέπει να συμβάλλει όπως το κάνει για την χρηματοπιστωτική εποπτεία για ένα φόρο επί των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο θέματα τα οποία ε, προασπίζουν την ανταγωνιστικότητα και τη θέση της ένωσης επίσης για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών των φορολογικών των μακροοικονομικών που πλήττουν την ένωση. Ε, για τον λόγο αυτό ε, ζητούμε οι επενδύσεις να έχουν μια οριζόντια διάσταση σε όλες τις πολιτικές της ένωσης και στην ατζέντα 2020. Ζητούμε μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επενδύσεις και μια σχετική ανακοίνωση, κύριε Επίτροπε, με δείκτες και παραμέτρους, όπως αυτή που επεξεργάζεται ο ΣΑ, ε, που θα αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες και θα μας βοηθούν να αποφασίσουμε για τις στοχευμένες παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε. δεν πρέπει να ε, ε, παραβλέπουμε ότι η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγορών ομολόγων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διεύρυνση της βάσης των επενδύσεων είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η επενδυτική πολιτική πρέπει να αποτελέσει βασικό εργαλείο και για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών βορρά και νότου δημοσιονομικών και άλλων ανισορροπιών. γι' αυτό μια ε, καινοτόμα πρόταση είναι η δημιουργία ενός ευρωπαρατηρητηρίου που θα παρακολουθεί τις τάσεις θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα ε, προτείνει πολιτικές ε, Προ την ενίσχυση την επενδυτική αλλά και επίσης για την προβολή της Ευρώπης ως επενδυτικού προορισμού στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε με το Catch the Έχουμε πάνω από πέντε αιτήματα. Θα δώσουμε το λόγο σε όσους δεν πήραν μέρος στην τελευταία συζήτηση. Ξεγερνάμε με τον κύριο Σεκέρσκι. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη είναι ένα σημαντικό σημείο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις και οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Προσπαθούν να βρουν ε, επενδυτές Πώς ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε την Ευρώπη ένα σημείο που αξίζει τον κόπο να επενδύσει κανείς. Η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη ρυθμίζεται πάρα πολύ καλά σε σχέση με άλλα μέρη στον κόσμο και η πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη εγγυάται στα σερές συνθήκες. Ε, ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η υψηλή ποιότητα των κεφαλαίων. Πού βρίσκεται λοιπόν το πρόβλημα. Πρόκειται για κοινωνικά υπεύθυνε υποθέσεις. Θα πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη του θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τις κοινωνικέ συνθήκες. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι ιδιαίτερα δαπανηρέ. Θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε και το, και το σύστημα το χρηματοπιστωτικό μα σύστημα. Αυτό συνδέεται με τη φορολογική πολιτική. Ευχαριστώ το λόγο κυρία, κυρία Ντάμψλα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το θέμα. Πρόσφατα γίναμε μάρτυρες διαμαρτυριών των εργαζομένων σε πολλά μέρη των εργαζομένων ήταν κατά της μετάταξης διάφορων εταιριών ε, εκτός της Ευρώπης. Το αποτέλεσμα είναι ότι δημιουργείται πάρα πολύ μεγάλη ανεργία. Για να αποφευχθούν αυτά στο μέλλον η Ευρώπη χρειάζεται μια στρατηγική προσέγγιση νέων και ξένων επενδυτών για να, διακρατική, για να προωθηθούν διακρατικές επενδύσεις αλλά και η μετακίνηση φοιτητών και εργαζομένων. Θα πρέπει να προωθήσουμε τη σύμπραξη δημόσιου και δικού τομέα, να στηρίξουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες και να τους δώσουμε πολλές ευκαιρίες. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις ε, ε, βιώσιμες επενδύσεις. Ο κύριος Πάσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συμφωνώ απόλυτα με τη δήλωση που υπάρχει στην έκθεση ότι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της Ένωσης σε σχέση με άλλες περιφέρειες είναι πάνω απ' όλα ο υψηλής μόρφωσης πληθυσμός, η τεχνική υψηλής, υψηλών προδιαγραφών υποδομή, και η τεχνολογική υποδομή που είναι πολύ προηγμένη. Πιστεύω ότι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ε, τα θέματα ενέργειας και η αυτονομία της σε αυτά τα θέματα. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε καινούρια θέματα που θα ξεπερνούν το έδαφος της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί, κατασκευαστές, φεύγουν από την Ευρώπη και πάνε στη Ρωσία, την Κίνα, τη Βραζιλία. Αυτό δείχνει ότι οι συνθήκες που προσφέρουμε στους Ευρωπαίους επενδυτές είναι χειρότερες από αυτές που προσφέρονται αλλού. κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να συγχαρώ την συνάδελφο κυρία Κράτσα για το έργο της. Η παγκόσμια οικονομία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση τώρα, αλλά υπάρχουν ακόμα βασικά εμπόδια για τη σταθεροποίηση της ελεύθερης αγοράς. Η Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τα δύναμα σημεία και να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει για να προσελκύσει επενδύσεις ε, γι' αυτό χρειάζονται ταχείες ε, μεταρρυθμίσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, επικεντρωνόμενοι στην εσωτερική αγορά και δίνοντας σημαντικά ωφέλη για τους επενδυτές. Έχουμε το της Ράσια Μοντάνα στη Ρουμανία ένα επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και θέσεις εργασίας σε μια πληγήσα περιοχή. Μπορεί επίσης να συμβάλλει και στην εθνική οικονομία. Όμως ε, επειδή δεν υπάρχει απόφαση υπέρ ή κατά του προγράμματος αυτού, χάνουν την υπομονή τους οι ξένοι επενδυτές. Και τώρα κυρία Κλέπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω ο Σκιώδης από τους σοσιαλιστές, την κυρία Κράτσα, για την έκθεση αυτή για την βελτίωση των επενδύσεων που είναι πολύ σημαντική σε περίοδους κρίσης. Χρειαζόμαστε κοινέ κατευθυντήριε γραμμέ. Θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε τι ιδέε μα. Θα πρέπει προφανώ να φροντίσουμε και να επενδύσουμε για θέσει εργασία για του νέου και να θέσουμε σαφεί στόχου για τι ευρωπαϊκέ περιφέρειε και κοινότητε. Στην τροπολογία μου τάσομαι υπέρ των νέων επενδύσεων στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής και σε σχέση με το περιφερειακό επίπεδο, γιατί εκεί βλέπω αναπτυξιακές δυνατότητες και είναι πολύ σημαντικό την πραγματική οικονομία στην Ευρώπη να τη χρηματοδοτήσουμε και χρειαζόμαστε καλύτερη πολιτική που θα προσελκύσει στην Ευρώπη παγκόσμιους επενδυτές. Ευχαριστώ. Να ζητήσω από τον Επίτροπο κύριο Κάλλας να κάνει τις καταλεκτικές παρατηρήσεις για τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οφείλω να ομολογήσω ότι το θέμα αυτό με αγγίζει βαθύτατα, διότι στο παρελθόν ήταν βασικό στοιχείο της οικονομικής μας πολιτικής να προσελκύσουμε άμεσες ξένες επενδύσεις στη δική μου χώρα όταν κατακτήσαμε την ανεξαρτησία μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την έκθεση αυτή για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ευρώπη και ευχαριστεί την κυρία Κράτσα Τσαγκαροπούλου για την ε, σκληρή της δουλειά. Ε, στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία πρέπει να δημιουργήσουμε τις σωστές προϋποθέσεις έτσι ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να παράγουν και να είναι ανταγωνιστικές στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον. Πράγματι, αναδύονται ε, διάφορες άλλες οικονομίες και αυτό εντείνει τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, αυτό προσφέρει και νέες ευκαιρίες ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των εμπορικών συμφωνιών ε, και των επενδύσεων. Οι άμεσες ξένες απαιτήσει είναι βασικό ε, στοιχείο για όλα αυτά. Εμείς υποδεχόμαστε άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ευρώπη που ε, ανέρχονται σε 225 δις ευρώ από τον υπόλοιπο κόσμο μόνο για το 2011. Ωστόσο, το μερίδιο το ευρωπαϊκό στις ξένες άμεσες επενδύσεις έχει μειωθεί στον υπόλοιπο κόσμο από το 45% το 2001 στο 20% το 2010. Αυτή η μεγάλη ε, πτώση έχει σημειωθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας, αλλά θα πρέπει ε, να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την καλή θέση που έχουμε ε, στη διεθνή σειρά κατάταξης και μπορούμε να μάθουμε ένας από τον άλλον για τις καλές πρακτικές προκειμένου να προσελκύσουμε επενδύσεις. Και γνωρίζουμε τι προσελκύει τις ε, άμεσες ξένες επενδύσεις ουσιαστικά ο βασικός λόγος για τον οποίο παραμένει ελκυστικός ο προορισμός η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το υψηλά καταρτισμένο εργασιακό δυναμικό, η μείωση των κανονιστικών ρυθμίσεων για την ε, έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης, η υψηλή ε, ποιότητα των διαφόρων υπηρεσιών που προωθούν τις επενδύσεις και ε, τα διάφορα μέτρα που εφαρμόζουμε στο πλαίσιο της εφαρμογής ε, των πολιτικών μας. Έχουμε ψηλή παραγωγικότητα και έχουμε υποδομές ε, στους τομείς της τεχνολογίας, της ε, πληροφορικής μεταξύ άλλων. Και χαίρομαι διότι στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η συγκήτρια αναφέρεται σε όλες αυτές τις πτυχές του ζητήματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράγματι προετοιμάζει, καταρτίζει μια ανακοίνωση για τη βιομηχανική πολιτική και για τα πιο σημαντικά προϊόντα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο από το 2010 και μετά. Θα συνεχίσουμε να σκούμε πιέσεις ώστε να υπάρξει το σωστό πλαίσιο για να απελευθερώσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία το δυναμικό της. Και μιλούμε για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, για τη βελτίωση της ενίας αγοράς, για τη βιομηχανική καινοτομία, για τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά από το ίδιο σημείο κίνηση, από το οποίο ξεκινά και η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εντοπίζει του ίδιου τομεί όπου θα πρέπει να αναλυφθεί δράση. Κάποιες από τις συγκεκριμένε προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικές. Ε, ε, διατυπώνται το αίτημα για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού ε, Παρατηρητηρίου, για τη βελτίωση της συνεργασίας σε νομοθετικό επίπεδο. Είναι σωστά πράγματα και έχει γίνει πολλή δουλειά τα τελευταία χρόνια. Ε, τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διεξάγει διαλόγους με τους βασικούς εταίρους μας, εμπορικούς μας εταίρους και έχει διοργανώσει πολλές ε, εκδηλώσεις για την ανταλλαγή ε, καλών και ορθών πρακτικών. καλωσορίζω γενικότερα την προσέγγιση της έκθεσης η οποία επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί τομείς για επικοδομητική συνεργασία. Χαίρομαι διότι ε, ξεκινήσαμε τη σημερινή ε, συνεδρίαση συζητώντας τον ευρωπαϊκό, ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο όπου είναι όντως ένας τομέας όπου θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε επενδύσεις. Επανειλημμένως έχουμε συζητήσει την ομοθετική πράξη για την ενιαία αγορά και θα συνεχίσουμε με τη συζήτηση για την επόμενη ε, πρόταση που είναι πολύ σημαντική ε, για την προσέλκυση των ξένων επενδύσεων. Όλα δηλαδή είναι στα χέρια μας, είναι στο χέρι μας να έχουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνω τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12.30. Προχωρούμε στην έκθεση του κυρίου Μίλοσλαβ Ράνσντορφ «Εμπορικές πτυχές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης».